Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 15 θα το εξετάσουμε πριν από το 14 και το 20 ε, μετά από τα 17 και 18. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις Αν όχι, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεν έχω ανακοινώσεις. Πάμε στο 3. Έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ε, τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 20ης και 21ης Νοεμβρίου του 2017 θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σημείο 4. που είναι η πρώτη μας ψηφοφορία. Ελπίζω ότι έχετε μαζί σας τις ηλεκτρονικές σας κάρτες που τις έχετε τοποθετήσει μέσα στη σχισμή. Αρχίζουμε με την έκθεση Σάγερ. So, amendment number has been... Η 7 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 1 και 8. Υπέρ. Mm -hmm. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ελέγξουμε. Τη 10. Ηλεκτρονικός. Maybe one more. Μία ακόμη φορά, κύριε Άντερσον. Δύο εκθέσει Σάιερ υπάρχουν. Ποια ψηφίζουμε τώρα κύριε Πρόεδρε. Α, ναι, συγγνώμη. 2016-039. Ο χώρος δικαιοσύνης. Αυτό ψηφίζουμε τώρα. 0399, συγγνώμη. 2016-0399. Εντάξει. Κάποιος δεν ψήφισε. Να κλείσω την ψηφοφορία. Ωραία, την κλείνω. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 και 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 και 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Uh, maybe we control that. Να την ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικώς. Uh, we control 18. Τη 18. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικώς. I end the vote. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται sorry. Ε, then... Ε, Πάμε τώρα στην τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος και πάλι. Ηλεκτρονικός. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο εκθεσής ε, στο σύνολό του ηλεκτρονικός. Uh, I the Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την απόφαση έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, ή ηλεκτρονικός και πάλι. I end Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. κεφάλι Λοιπόν, υπάρχουν μία-δύο επιπλέον κάρτες ψηφοφορία ε, από τους παρισταμένους, σε σχέση με τους παρισταμένους, σας το λέω αυτό. Δεύτερη τώρα έκθεση Σάιερ, κα, καταρχάς σας συγχαρώ για την πρώτη έκθεση, τον κύριο Σάιερ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δεύτερη που είναι πολύ μακροσκελέστερη. Τροπολογία 1 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 94. Στη σελίδα 14. Δεν είναι και πολύ οικολογικό αυτό. Έχετε όλη την τροπολογία 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 177 που είναι στη σελίδα 25. Για κάποιους είναι 23 η σελίδα. 177. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 και 595 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πάμε στην τροπολογία 388 στη σελίδα 51 όχι για όλους όμως την ίδια σελίδα This one? Yes. Everybody has three... Εντάξει, βρήκατε την 388. Ωραία, υπέρ. Κατά. Ε, τότε να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς καλύτερα αυτήν την τροπολογία. Πέρας εγκρίνεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 391 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 392 και 393 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο έκθεση στο σύνολό του, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας, εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο ηλεκτρονικός επίσης. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. Συγχαρητήρια και πάλι κύριε Σάιερ. Now, Αυτό ήταν λοιπόν η προθέρμανση και τώρα περνάμε στην έκθεση Χαουταλά και ορισμένες πτυχές που αφορούν ε, τις ε, συμβάσεις για πωλήσει αγαθών. Τροπολογία 41 είναι η πρώτη, υπέρ, κατά, αποχές, ε, παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ένα υπέρ. Αλέχος. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ αποχές εγώ θα λέγω ότι απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ εγκρίνεται 119 υπέρ 119 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται Εκατόν υπέρ κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Yes. It has been adopted. Μάλιστα, εγκρίθηκε. 245 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά κύριε Φώσο. Τον κατάλογο ψηφοφορίας λέει ότι καταπίπτει εάν η συμβιβαστική 1 εγκριθεί. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν εγκρίθηκε, απορρίφθηκε. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Μάλιστα. Θα αναψηφίζουμε 126 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε άλλη μια φορά παρακαλώ ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. 120, ε, 22 ε, in favor. 22 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ Εγώ στις σημειώσεις μου λέει ότι μετά τη συμβιβαστική, εάν εγκριθεί, πάμε στην 136. Ναι. Λοιπόν, 136 ψηφίζουμε υπέρ. Against. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. not the hand, you I don't see. Yeah. And it has been rejected. Απορρίφθηκε. 251 in favor. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Για 251. Rejected. Απορρίφθηκε. Την ίδια πλειοψηφία έχουμε. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχέσε απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 153. Υπέρ κατά Να ελέγξουμε παρακαλώ 153. Απορρίφθηκε. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Για την 21. Εγώ από εδώ που σας βλέπω μου φαίνεται σαφές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, λάθος έκανα. Υπέρ της 156. Κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε παρακαλώ. εγκρίνεται. 157 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, λάθος. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, έλεγχος ηλεκτρονικός. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Maybe, but... This has been rejected. Um, Then we go 161 in favor. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. 171 υπέρ κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 171 yes. Rejected. Uh, Απορρίφθηκε. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Α, έχει καταπέσει. Α, τότε δικό μου λάθος. Η 176 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Απορρίφθηκε. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τι θέλετε να ελέγξουμε ωραία να ελέγξουμε για την συμβιβαστική 8 Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά να ελέγξουμε τα 207 παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Διακόσια δύο υπέρ. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές ε, γίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για τις 45 εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 καταπίπτει. 217 δεκαεπτά υπέρ καλά κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά να ελέγξουμε Ελέγχουμε την 49. Εγκρίθηκε. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 καταπίπτει Οι δύο υπέρ κατά Α, υπάρχουν δύο τμήματα μάλιστα το πρώτο τμήμα χωρίς το τμήμα που λέει όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο γίνεται. Υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ Πέντα εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται We just voted 64. Μόλις ψηφίσαμε την 64. Εγκρίθηκε και πάμε στην 65, εντάξει. Η 251 δεν εγκρίθηκε, απορρίφθηκε. Άρα λοιπόν η 67 έχει καταπέσει. Η 251 απορρίφθηκε και γι' αυτό το λόγο η 251 δεν εγκρίθηκε και γι' αυτό το λόγο και η 67 ε, καταπίπτει. Είμαστε στα 65 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 όχι συγγνώμη λέει ο πρόεδρος 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά ελέγχουμε για την 74 εγκρίνεται 2.31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 77 απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.33 υπέρ κατά να ελέγξουμε για τη 233 απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 ναι, να ελέγξουμε το 235 ε, ε, ψηφίστε απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά δεν είμαι βεβαία Έλεγχος για την 87. Απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά δεν θα πρέπει να ελέγξω απορρίπτεται 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Yes. 239 uh, in favor. 239 υπέρ Now, May I check then on two... Να ελέγξουμε για το 239. It has been rejected. Απορρίφθηκε. Then amendment 6 that falls. Uh... Τροπολογία 6 καταπίπτει. 97 in favor. 97 again. 97 υπέρ λοιπόν κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εγώ λέω ότι απορρίπτεται αλλά σε ελέγξουμε. Yeah. Rejected. Uh... Απορρίφθηκε. 101. Yes. 101 in favor. 101 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές ε, γκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται yeah. 105 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 240 in favor υπέρ κατά ε, της εκατόν... ε, ε, νέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, συγγνώμη εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε Α, εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 242 υπέρ κατά αποχές ε, απορριπτήκε 113 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 114 Όχι, 113. 113 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Τώρα, ολόκληρο το σχέδιο γνωμοδότησης, ηλεκτρονικά Απορρίφθηκε. So, now I cannot say... Τι να πω, συγχαρητήρια στον κύριο Σάιερ. Δεν μπορώ. Α, όχι, με συγχωρείτε στην κυρία Χάουταλα. Χάουταλα, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Now we are voting on... Θα ψηφίσουμε τώρα συνεχίζει ο πρόεδρο τη δική μου γνωμοδότηση. Πρόκειται για την απαλλαγή. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Κυρία Γκέπχαρτ, εσείς. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να δηλώσω για ποιο λόγο η πολιτική μου ομάδα κατεψήφισε τη γνωμοδότηση. Το τελικό κείμενο όπως προέκυψε από την ψηφοφορία, αποτελεί κείμενο το οποίο αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών και καταναλωτριών σε πολλές χώρες μεταξύ αυτών και τη Μεγάλη Βρετανία αλλά δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ τα μειώνει τα δικαιώματα των καταναλωτριών και καταναλωτών και δεν μπορούμε να δεχτούμε δικαιώματα των πολιτών να καταργούνται μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου. Και αυτό για μένα είναι απόλυτη ξεδιαντροπιά. Αυτό ψηφίστηκε εδώ. Και γι' αυτό χαίρομαι που εν τέλει απορρίφθηκε το σύνολο της γνωμοδοτήσεω. Βέβαια τώρα το ερώτημα που θέτω προ εσά, κύριε Πρόεδρε είναι το εξή. Βρισκόμαστε στην διαδικασία του άρθρου 54. Ποια είναι η συνέχεια τώρα? Διότι δεν έχουμε γνωμοδότηση προς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή παρόλο που έχουμε διαδικασία του άρθρου 54. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, μπορείτε να με ενημερώσετε. και Κύριε Χάουταλα, ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από τα επιχειρήματα των σοσιαλιστών δημοκρατών που εκφράστηκαν μόλις τώρα μετά από την απόρριψη τη γνωμοδότηση της οποίας υπήρξα συντάκτρια. Πιστεύω επίσης όμως, οφείλω να ομολογήσω, ότι ως νομική επιτροπή έχουμε καταλήξει σε μια κατάσταση όπου συχνά, πολύ συχνά είμαστε διασπασμένοι. Δεν έχουμε ξεκάθαρες ή μάλλον δεν έχουμε στέρεες πλειοψηφίες. Πότε κινείται από τη μια, πότε από την άλλη. Ούτε βλέπω άλλωστε, αυτό είναι ατυχέ, ούτε βλέπω άλλωστε να εκπροσωπούνται πραγματικά όλε οι πολιτικέ ομάδε. Εγώ δεν αποσύρω το όνομά μου, όμω είμαι και εγώ πολύ περίεργη σχετικά με το ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας άρθρου 54 και της συμμετοχής της, νομική της Νομικής Επιτροπής μάλλον στις ε, περαιτέρω διαβουλεύσεις. The rules of Ο κανονισμός δεν λέει τίποτα σχετικά. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση που προσωμιάζει με μια κατάσταση όπου δεν θα δώσουμε γνωμοδότηση, σαν δηλαδή να μην έχουμε ζητήσει εφαρμογή του άρθρου 54. Αυτό είναι η απάντησή μου. Επανέρχομαι στην ε, ψηφοφορία, στις ψηφοφορίες μάλλον καλύτερα. Η δική μου τώρα γνωμοδότηση για την απαλλαγή που αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά. Παρακαλώ να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 2. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3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 αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά παρακαλώ επαλήθευση απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ επαλήθευση 19 εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά παρακαλώ επαλήθευση 27 εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στο σύνολό της η γνωμοδότηση παρακαλώ ηλεκτρονικά εγκρίνεται. Ας συγχαρώ τον εαυτό μου λοιπόν και η τελική ψηφοφορία, η τελευταία μάλλον, είναι για την γνωμοδότηση για την νομική βάση, γνωμοδότηση του κυρίου Άξελ Φως. Μπορούμε να ψηφίσουμε και με ανάταση των χεριών. Υπέρ, α, όχι με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λάθος μου, ηλεκτρονικός Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Βόση. Τέλος των ψηφοφοριών. Τώρα θα συνεχίσουμε στις 11 η ώρα με κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών νομικών και συνταγματικών. Παρακαλείστε να περιμένετε λίγο.